Okay, colleagues, we're going now to... Περνάμε τώρα στο σημείο 21, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο είναι... Η εκρόση είναι από κοινού με την Επιτροπή ΦΑΝ. Θα μιλήσουμε για, το, για την πρωτοβουλία Spotlight μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλληψη της βίας ενάντια στις γυναίκες και στα νερά κορίτσια. Έχουμε μαζί μας την Επίτροπο Μίμικα, η οποία από τη στιγμή, ο οποίος από τη στιγμή που ανέλαβε το ρόλο του ως επίτροπος, ο επίτροπος Μιμίτσα, ανέλαβε ότι ε, ε, δεσμεύτηκε στο ότι θα είναι μια φεμινιστική επιτροπή. Έχουμε και την κυρία Αλκέτα Ξάφα Μυρίπα, η οποία είναι μια ακτιβίστρια και conceptual καλλιτέχνηδα. Βεβαίως αυτή είναι η εβδομάδα δράσεις για τα νεαρά κορίτσια. Σήμερα είχαμε στο Κοινοβούλιο επισκέπτες γυναίκες που σήμερα εμένα ε, μου πήραν συνέντευξη. Συζητήσαμε για το ότι δεν θα πρέπει απλά να μένουμε στην θεωρία, αλλά να περάσουμε στην πράξη και βεβαίως στις 11 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα a Girl Child. Θα μιλήσουμε για την πρωτοβουλία, όπως είπαμε, Spotlight για την εξάλληψη της βίας ενάντια στις γυναίκες και στα νεαρά κορίτσια. Ένας ακόμη λόγος που είμαι χαρούμενη σήμερα είναι γιατί, όπως όλοι γνωρίζετε, η Επιτροπή Νόμπελ έδωσε στην Άντια Μουράτ και στον dr. Μαγκουέγγι με το, το Νόμπελ Ειρήνης στα δύο αυτά άτομα που εδώ και χρόνια δουλεύουν, εργάζονται για την εξάλληψη της βίας, για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Η Νάντια Μουράν, την οποία κανείς μας πιστεύω δεν θα ξεχάσει τους λόγους της, τις δικές μας ολομέλειες εδώ στο Κοινοβούλιο, όταν μας εξήγησε πώς και η ίδια είχε βρεθεί, την είχαν απαγάγει και ε, μοιράστηκε μαζί, της, μαζί μας τις δικές της εμπειρίες κατά τη διάρκεια της α, κράτησής της. Α, το γεγονός ότι απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης μας δείχνει ότι η Επιτροπή για την απονομή των Νόμπελ λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τα ζητήματα αυτά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την πρωτοβουλία Spotlight που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 με 500 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Το σκεπτικό είναι να επενδύσουμε σε προγράμματα για την καταπολέμηση της, για την εξάλληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και για την καταπολέμηση της βίας ενάντια στις γυναίκες. Θα έχουμε δύο, θα είναι, θα, η συνεδρίαση μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Πρώτα έχουμε την παρουσίαση του Επιτρόπου και στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση και μετά θα έχουμε την παρουσίαση της ΜΡΙΠΑ. Θέλω λίγο να δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου Βίλια Μπλίνκεβίτσουτε το όνομά της είναι κάπως πολύπλοκο να το προφέρω Είναι πρόεδρος της Επιτροπής ΦΑΜ και είναι χαρά μας να την καλωσορίσουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω κι εγώ τη Λίντα, τον Επίτροπο. Βράτομαι τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΔΕΒΕ για την άριστη συνεργασία. Καθότι μας ενδιαφέρουν, α, έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. όλοι γνωρίζουμε την έκταση που έχει βία ενάντια στις γυναίκες στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο, μία στις πέντε γυναίκες, τουλάχιστον μία φορά και τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους, αντιμετωπίζει περιστατικά βίας εναντίον τους. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει, θα πρέπει να καταψηφίσει το ώστε να δώσει εργαλεία στις γυναίκες για να καταπολεμήσουν αυτού του τύπου τη βία. Κάτι τέτοιο επιχειρεί η πρωτοβουλία Spotlight. Είναι πολύ χρήσιμο να δούμε σε τι φάση βρίσκεται η επιλογή της, η εφαρμογή με της πρωτοβουλίας αυτής που διανύει τον πρώτο χρόνο της ζωής της. Χαίρομαι που, έχω μας, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Επίτροπος Μίμητσα και η κυρία Μρίρα για να κάνει την παρουσίασή της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρωση λοιπόν να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Μίμητσα. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές πρόεδροι, αγαπητά μέλη, συνάδελφοι και φίλοι. Σας ευχαριστώ όπως πάντα για το θερμό καλωσόρισμά σας και από τις δύο επιτροπές. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε και επίσης ε, στην έμφαση που θα δώσουμε στην πρωτοβουλία Spotlight. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δούμε πώς θα πήγαμε σε αυτό το πρώτο χρόνο της ζωής μας και να δούμε και ποια είναι τα σχέδιά μας για, ε, για το χρόνο που έρχεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη, εκπροσωπώντας τις καθολικές ε, μας αξίες, τις παγκόσμιες αξίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, αποφάσισε να ενδυναμώσει τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και την συνεργασία μας ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Αποκινούμε τον ε, Γενικό Γραμματέα Μιλ Μοχάμεντ, εκδώσαμε μία δήλωση όπου περιγράψαμε πώς θα ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας. Και σε μια, περίοδο, που οι συνεργασίες δεν ε, ε, ευδοκιμούν. Πρακτικά, πώς θα το καταφέρουμε λοιπόν αυτό. Μα θα πρέπει να μοιραστούμε τις γνώσεις μας ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μία από τις πιο κατάφορες ε, παραβιάσεις των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έθραυσα μέλη της κοινωνίας, οι γυναίκες, κορίτσια βλέπουν τα δικαιώματά τους να παραβιάζονται. Οικοδομώντας λοιπόν πάνω σε πρακτικές που γνωρίζουμε, η πρωτοβουλία Spotlight αναφέρεται σε μορφές βίας στην Καραϊβική, στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική και προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις πολιτικές ε, προσπαθούμε να αλλάξουμε ζωές και προσπαθούμε να αλλάξουμε και νοοτροπίες. Η αρχική μας επένδυση των 500 εκατομμυρίων ευρώ είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχουμε κάνει για τέτοιου τύπου σκοπό. Ήταν μια προσωπική μου δέσμευση, αλλά ήταν και μια υπόσχεση που έδωσα σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Να εξασφαλίσω ότι οι πράξεις μας για να ενδυναμώσουμε και να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα ναρά κορίτσια δεν θα παραμείνουν λόγια και ευχές. Θα στηρίξουμε τους στόχους μας αυτούς με πράξεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ είναι μια πραγματική όθηση, ούτω ώστε να προωθήσουμε την παγκόσμια δράση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ισπανία που έχουν ήδη δηλώσει έμπρακτα τη στήριξή τους σε αυτήν την πρωτοβουλία. Το προηγούμενο Νοέμβριο ανακοινώσαμε το πρώτο περιφερειακό πρόγραμμα στην Ασία για να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες μετανάστες που, που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της περιοχής από ακτιβίστριες στην Μπαγκόκ που προσπαθούν να δώσουν φωνή σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλες αυτές τις γυναίκες που δεν ε, μπορούν να έχουν μια δίωδο επικοινωνίας. Το προηγούμενο μήνα στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσα και το δεύτερο περιφερειακό μας πρόγραμμα για την Λατινική Αμερική σε ό,τι αφορά τις δολοφονίες γυναικών. 12 γυναίκες δολοφονούνται στην περιοχή αυτή κάθε μέρα. 98% από αυτές τις δολοφονίες δεν διώκονται ποτέ πινακά και αυτό απλούστατα δεν είναι αποδεκτό. 50, τα 50 εκατομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν προς αυτό το πρόγραμμα θα επικεντρωθούν στις πέντε χώρες που έχουν τα, μεγαλύτερα, περισσότερα θύματα. Αλτζεντίνα, Ελσαρβαντόρ, Χοντούρα, Γκουατεμάλα και Μεξικό. Θα μας επιτρέψουν επίσης να α, χτίσουμε στην πολιτική μας θέληση να σταματήσουν οι δολοφονίες γυναικών, κάτι που στηρίζεται από όλε τις κυβερνήσεις. Στην παρουσίαση του προγράμματος αυτών είχα την τιμή να συνοδεύομαι από πάρα πολλές άξιες γυναίκες και να ακούσω τη μαρτυρία της Νατάλια Πομφρέντε Λεόν, η οποία συγκίνησε το ακροατήριο. Ήταν ένα από τα πολλά θύματα α, επίθεσης με οξύ στην Κολομβία, κάτι το οποίο στη χώρα εκείνη θεωρείται ένα απλό αδίκημα η φρικτή αυτή πράξη που δεν αναγνωρίζεται και δεν τιμωρείται, τώρα πλέον αντιμετωπίζεται με ένα νόμο που φέρει το όνομά της. Η Νατάλια εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που αποτελεί πρωτοβουλία αυτό. Γυναίκες που αρνούνται να σιωπήσουν μέχρι ότου όλοι οι πολίτες ζουν σε έναν κόσμο χωρίς φόβο την ε, θέλησή μας να ρίξουμε φως σε μερικά από τα πιο ε, σκοτεινά σημεία του πλανήτη αυτού, του κόσμου αυτού. Θα αναφερθώ στο φαινόμενο της πεταλούδας, γιατί ξέρω ότι κάθε γυναίκα και νεαρό κορίτσι μπορεί να έχει τη δύναμη ενός τυφώνα, αν απλώς μπορέσει να απλώσει τα φτερά της. Και αυτό θα πρέπει να τους βοηθάει να κάνουν αυτή η πρωτοβουλία Spotlight. Το πρόγραμμα για την Αφρική θα πρέπει να ξεκινήσει πριν το τέλος του χρόνου και στις αρχές του επόμενου χρόνου τα προγράμματα για την Καραϊβική. Κυρίες και κύριοι, πριν ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, επιτρέψτε μου απλά να σας πω πόσο σημαντικό είναι το spotlight σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στην δική σας στήριξη και χάρη στην βοήθειά σας, πάντοτε στηρίζει την ισότητα των δύο φύλων. Αλλά ποτέ δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε επιτύχει τους στόχους μας μέχρι ότου κάθε γυναίκα και κάθε νερό κορίτσι ζει σε συνθήκες ασφάλειας τα δεδομένα που έχουμε είναι πραγματικά σοκαριστικά. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Το σχέδιο δράσης μας για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων έχει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για να μπορέσει να αλλάξει τις ζωές των γυναικών και των νέων κοριτσιών σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές θα μπορέσουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη δεύτερη αναφορά πρόοδου που με μεγάλη περηφάνεια σας λέω ότι πραγματικά κάνει τη διαφορά. Υπάρχει μια τεράστια αύξηση στον αριθμό δραστηριοτήτων που λαμβάνουν πολλές ε, χώρες για την ισότητα των δύο φύλων περισσότερο από το 65% την προηγούμενη χρονιά σε σχέση με το 47% για το 2015 έχει να κάνει με την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Είμαστε λοιπόν σε καλό δρόμο. Στόχος μας είναι το 85% των συνολικών επενδύσεων να προωθεί την ισότητα των δύο φύλων μέχρι το 2020. Κυρίες και κύριοι, η ανακοίνωση των ε, νικητών του Νόμπελ Ειρήνης την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ε, μια συγκινητική στιγμή για όλους μας εδώ, για όλους εμάς αυτό το δωμάτιο. Να δούμε ότι οι θυσίες της Νάντια Μουράτ και του Ντάνεξ Μακουέγγι αναγνωρίστηκαν είναι κάτι που εμένα προσωπικά μου δίνει ελπίδα. Και με κάνει να πιστεύω ότι είναι δυνατό το τέλος της βίας ενάντια στις γυναίκες πριν το τέλος της δικής μας γενιάς. Θα πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα λοιπόν για να δούμε την πρωτοβουλία Spotlight να αναπτύσσεται σε κάθε περιοχή και να αλλάζει τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών για το καλύτερο. Σε αυτήν και σε όλες μας τις προσπάθειες εξακολουθούμε να βασιζόμαστε στη δική σας στήριξη, στις δικές σας εμπειρίες και στην δέσμευσή σας στο σκοπό μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την προσοχή σας και ανυπομονώ να ακούσω τις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας αλλά και την συμβολή σας όχι μόνο στην καταπολέμηση της βίας αναντίον των γυναικών, αλλά και σε όλες τις δράσεις μας που αφορούν στην ισότητα των δύο φίλων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για την ισχυρή του δέσμευση για αυτό το θέμα, στο οποίο βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος επί τόπου. Έχουμε τις ερωτήσεις σε δύο τμήματα, Πεσέρα και μετά Χάιντι Χάουταλα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε γιατί βρίσκεστε εδώ σήμερα σε μια χρονική στιγμή γλυκόπικρη θα έλεγα διότι από τη μία πλευρά είναι καταπληκτικά τα νέα σύμφωνα με τα οποία οι δικοί μας υποψήφοι έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την αταλάντευτη μάχη τους για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών, ε, τη χρήση ε, της βίας ως όπλο πολέμου. Θα πρέπει να συγχαρούμε θερμά αυτούς τους δύο υποψηφίους μας, αλλά και τους εαυτούς μας ε, για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Είχαμε συμφωνία με αυτούς από το 2014 και το 2016. Το βραβείο Ζαχάροφ μας, μας δεσμεύει φόρου ζωής. Είναι το πιο προφανές όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υποχρέωσή μας όλες τις προσπάθειες και όλους τους πόρους μας να τους στρέψουμε ε, ε, έτσι ώστε να τους πλαισιώσουμε σε αυτόν τον αγώνα για την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτή είναι και η περίπτωση της Νάντια Μουράτ η οποία συνεχίζει να λέει ότι όσοι έχουν διαπράξει αυτή τη γενοκτονία και αυτό τον υπέρμετρο είναι υπόλογοι για αυτό τον υπέρμετρο τρόμο που έχουν σπείρει θα πρέπει να απολογηθούν ενώπιον των ε, αρμοδίων αρχών. Όλοι λοιπόν έχουμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση και μας προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν ακυρώσει ακόμα τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι το πιο εμπεριστατωμένο, το πιο άρτιο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς η Πολωνία μάλιστα απειλεί ότι θα αποσύρει την υπογραφή της από την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και άλλες χώρες έχουν απειλήσει ότι θα οπισθοχωρήσουν και θα αποσυρθούν. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην κυρώσει τη σύμβαση αυτή ως οντότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και χρειάζεται να το πράξουν και οι χώρες η κάθε μία ξεχωριστά. Γιατί αυτό αντιστοιχεί, αυτό περιμένουν από εμά από τη στιγμή που είμαστε νομοθέτης, να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Η πρωτοβουλία Spotlight είναι ε, ένα από τα καλύτερα νέα που έχουμε να κομίσουμε για την ατζέντα του 2000 και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε Έχουμε τους στόχους μας με συγκεκριμένες ημερομηνίες, με συγκεκριμένους στόχους και με πόρους και χρήματα που θα στηρίξουν ε, τους στόχους έτσι ώστε αυτοί να μην παραμείνουν στο επίπεδο των ε, ε, ηθικών και καλών προθέσεων και να μην παραμείνουν στη σφαίρα του θεωρητικού, για να δοθεί ένα τέλος πια στη βία εναντίον κοριτσιών και γυναικών σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει για να επιτευχθούν όλα αυτά να γίνουν και οι απαραίτητε αλλαγέ στο πολιτιστικό επίπεδο, στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Να εμπλέκονται τα μικρά αγόρια και κορίτσια από νωρί σε αυτή τη διαδικασία, στα πρώτα βήματα που κάνουν στον κόσμο μα, να καταλαβαίνουν ε, πώ ε, πρέπει να προχωρήσουν. Είμαστε σε μια στιγμή σιγουριάς και οπτικοποίησης, ε, μια στιγμή η οποία είναι πρωτοφανή σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι το οποίο το συνηθισμένο για αιώνες, δεν είναι πια συνηθισμένο και δεν είναι πια αποδεκτό και αυτό είναι κάτι που ξέρουμε και πιστεύουμε και προσυπογράφουμε όλοι. Αυτό το μήνυμα λοιπόν το Spotlight για την Λατινική Αμερική είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αποκτήσει περισσότερη σάρκα και οστά. Αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να αξιοποιηθούν με το σωστό τρόπο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε έναν κόσμο δίκαιο όπου θα συμβιώνουμε ειρηνικά και αρμονικά χωρίς να απελευθερώσουμε τις γυναίκες από τη σεξουαλική και άλλη βία την οποία υφίστανται. Ευχαριστώ θερμά τον Επίτροπο και ε, δηλώνω την ετοιμότητά μου να συμβάλλω με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι και η Νάντια Μουράτ και ο γιατρός ο Δόκτωρ Κουέγκε, οι δύο ε, στους οποίους απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, πράγματι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικές οι προσπάθειές τους. Σας ευχαριστούμε που μας τα θυμήσατε όλα αυτά. Η Χάιντε Χάουταλα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την ομιλία του, που ήταν πολύ εμπνευσμένη και κατάφερε να εμπνεύσει και εμά για την πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο κοινοβουλευτικό μας έργο. Η Βεατρίκη εξήγησε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν ζητήματα και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και οφείλουμε να υιοθετήσουμε μια μόνιμη δράση συγκεκριμένη έτσι ώστε να μην οπισθοχωρήσουμε σε σχέση με τα επιτεύγματά μας. Αναφερθήκατε στην τρομακτική ασυλία και ατιμεωρησία που επικρατεί στη Λατινική Αμερική. Οι χώρες που αναφέρονται, η, Ονδούρες, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, η Αργεντινή, το Ελσαλβαδόρ, εξ όσων γνωρίζω, είναι και χώρες όπου έχουν, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, ε, οι πιο ισχυροί περιορισμοί στο δικαίωμα της άμβλωσης, στο δικαίωμα της άμβλωσης σε ασφαλείς συνθήκες. Λοιπόν, ε, ε, θεωρείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο. Μπορεί η πρωτοβουλία Spotlight να βοηθήσει αυτές τις χώρες να καταλάβουν το εξή απλό, ότι δηλαδή αν θέλουν να μειώσουν την οδύνη και τα προβλήματα των παράνομων αμβλώσεων και τα προβλήματα υγείας και διάφορα άλλα για τις γυναίκες, τις οικογένειες και την κοινωνία, τότε θα πρέπει να έχουν πιο προοδευτική νομοθεσία. Και μετά, δεύτερο ερώτημα για τους γάμους με παιδιά είναι αυτό το πεδίο εφαρμογή ε, τη πολιτική σας. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει αυτό το γάμο με παιδιά που αποτελεί κατάφορη παραβίαση και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάφορο πλήγμα σε μια αξιοπρεπή ζωή ε, για τα νεαρά κορίτσια και αγόρια βεβαίω, αλλά τα κορίτσια είναι πολύ περισσότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά. Ευχαριστώ η Julie Ward παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, διότι ήρθατε να μας επισκεφτείτε, χαίρομαι διότι οι δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν από κοινού για μια εξαιρετικά σημαντική κατά τη γνώμη μου συζήτηση. Συμμερίζομαι απολύτως τα σχόλια των προηγούμενων συναδέλφων. Ξέρετε, ήμουν εκπρόσωπος του UNCSW, ε, ε, στο UNCSW, το Μάρτιο στη Νέα Υόρκη και τα δύο προηγούμενα χρόνια είχα πάει και εντωμεταξύ έχουν σημειωθεί ριζοσπαστικέ αλλαγέ σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση που υιοθετούν οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Και αυτό άλλαξε πλήρω τον τόνο των συζητήσεων ε, σε σχέση με δύο χρόνια πριν στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, Προηγουμένως, παλαιότερα, δύο χρόνια πριν, είχαμε αγωνιστεί να χτίσουμε γέφυρες με αφρικανικές οργανώσεις, με τους εταίρους μας, με ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, μεταξύ άλλων. Το Μάρτιο φέτος, οι ίδιοι άνθρωποι και αυτές οι οργανώσεις ε, ε, ήταν στο πλευρό μας, οι ίδιες από μόνο τους συμπαρατάχθηκαν με εμάς εξ αρχής, γιατί συνειδητοποίησαν ότι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, η υπερδύναμη, η μέγιστη, δεν είναι πια φίλη χώρα των γυναικών. Μόλις ε, ε, επιστρέψατε μόλις από τη Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι. Έχετε μπει σε αυτό το κλίμα, έχετε συνομιλήσει με τους διεθνείς εταίρους μας. Μπορείτε να μας δώσετε μια αίσθηση ε, του πού βρισκόμαστε από πολιτική σκοπιάς. Οι Αφρικανοί εταίροι ε, ε, συμπορεύονται μαζί μας, συνεχίζουν να, πορευ... να θέλουν να πορευτούν δίπλα μας. Ε, ποια είναι η συμβουλή σας, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τις γέφυρες που έχουμε χτίσει, πώς μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε τις αξίες μας και να συνεργαστούμε από κοινού. Γιατί έχουμε και τη Σύνοδο των Χωρών ΑΚΕ και πολλοί από εμά, ε, ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε χαρτοφυλάκια και αρμοδιότητε και για αυτά τα θέματα τη Αφρική, αλλά και για τι τις χώρες ΑΚΕ γενικότερο. Ε, και είναι θέματα διασταυρούμενα, αν θέλετε, που διασχίζουν εγκάρσια και αφορούν διάφορε γεωγραφικέ περιοχέ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχύσουμε ε, τι σχέσει αυτέ. Η Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο Επίτροπος παρακαλώ να απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ναι. Σας ευχαριστώ καταρχάς κύριε, και κύριοι βουλευτές για την στήριξη των δράσεων μας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Παράδειγμα κοινή δράσης και δέσμευση ισχυρής για να πετύχουμε τους στόχους αυτών των πρωτοβουλειών. Υπάρχουν κάποια επιμέρους ζητήματα που πηγαίνουν πέρα αυτής της πρωτοβουλίας Spotlight. Καταρχάς να σας πω ότι αυτή η πρωτοβουλία ως πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και είναι μια ευρία έννοια. στα προγράμματα μας στο μοθετικό πλαίσιο και στις προϊκές δράσεις να αλλάξουμε τις νοοτροπίες. Θα θέλαμε λοιπόν να επικεντρωθούμε σε όλες τις πτυχές της, γεία, της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Αυτές οι μορφές βίας είναι πολύ ευρείες αν σε μια γυναίκα αποτρέπεται ή απαγορεύεται η πρόσβαση στην απαγορευτική υγεία ή δεν της επιτρέπεται ή περιορίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, στον οικογενειακό σχεδιασμό. Και αυτά είναι μορφές βίας κατά τους. Δεν θέλουμε λοιπόν να είμαστε περιορισμένοι. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε όλες, όσο πιο πολλές πτυχές γίνεται της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και αυτό βεβαίω μας κάνει να αναρωτιόμαστε για το ρόλο της Ένωσης ως ανταπόκριση και στις αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης για την επαναφορά της πολιτικής τους με το Μεξικό. Γιατί θεωρούμε ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής δεν είναι καλό νέο για τις φτωχότερες γυναίκες του κόσμου. Οι αναπορικές υπηρεσίες υγείας και ο οικογενειακός σχεδιασμός παρουσιάζουν κάποιες επιπλοκές και έχουν σχέση όλα αυτά με τη θνησιμότητα, με τους, ε, με τους, τους και θα οδηγήσει σε περισσότερες αμβλώσεις πολλές από τις οποίες ε, γίνονται υπό ανασφαλείς συνθήκες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση ώστε να αντισταθμίσουμε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Όπως ξέρετε η Κομισιόν σέβεται την αυτονομία των χωρών εταίρων να αποφασίσουν όπως επιθυμούν για αυτά τα θέματα, αυλώσεις κλπ. και δεν επιβάλλει περιορισμούς στα πλαίσια των πολιτικών βοήθειας για την ανάπτυξη. Οπότε για εμάς οι δεν είναι όργανο ή εργαλείο οικογενειακού σχεδιασμού. Εμείς θεωρούμε να θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας στις χώρες εταίρους μας, ώστε να επιτρέψουμε στα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν αυτές τις παρεμβάσεις που προβλέπονται ως παρεμβάσει από τις πολιτικές προτεραιότητες, τι εθνικέ. Με αυτή λοιπόν την πρωτοβουλία μας, Spotlight, με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ αντιμετωπίζουμε τα θέματα του οικογενειακού σχεδιασμού και την αντισύλληψη όχι ως αντιμετώπιση της προσέγγισης της κυβέρνησης των τον είπα και των αποφάσεών της, γιατί ξέρετε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος φορέας παροχής βοήθειας για την ανάπτυξη. Οπότε οι δράσεις μας τωρινές για την ανάπτυξη θα καθοριστούν από τη δική μας ευθύνη και τη δική μας αλληλεγγύη. Επειδή, όπως είπα και ξαναλέω, είμαστε ο μεγαλύτερος πάροχος αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Και όλα αυτά ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν οι άλλοι σε αυτό το τομέα. Και αυτό λοιπόν θα αποτελέσει τμήμα της πρωτοβουλίας μας. Οικογενειακός σχεδιασμό, δικαιώματα και υγεία αναπαραγωγική και πρόσβαση, αντισύλληψη και προγράμματα αντισύλληψης. Αυτά είναι για μας σημαντικό τμήμα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Για τους γάμους, νομίζω ότι προσαρμοζόμαστε περιφερειακά και η καταναγκαστικοί γάμοι των παιδιών θα αντιμετωπιστούν μέσω κυρίως του αφρικανικού μας προγράμματος που υπογράψαμε με τον ΟΗΕ και θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα με το ίμιση από το σύνολο των 500 εκατομμυρίων του Spotlight. ώστε να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων και των καταναστικών γάμων των κοριτσιών. Επίσης, τονίσαμε σήμερα και τη σημασία της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης Η σύμβαση αυτή είναι το πρώτο διεθνές εργαλείο για τη θέσπιση νομικώς δεσμευτικών προδιαγραφών και προτύπων για να προστατεύσουμε τα θύματα και να τιμωρήσουμε τους θύτες. Όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης επέγραψαν αυτή τη σύμβαση, όπως και η Ένωση στο σύνολό της. Η επικύρωση λοιπόν της σύμβασης και σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο είναι κάτι κρίσιμη σημασίας. Η Κομισιόν συνεχίζει να καλεί τις χώρες μέλη να επικυρώσουν τη συμφωνία αυτή, τη σύμβαση αυτή, το ταχύτερο δυνατό και συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης ώστε να μεταφέρουμε θετικά μηνύματα σε σχέση με τα ωφέλη της σύμβασης. Και το κάνουμε όποτε μπορούμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ για την δέσμευσή σας που είναι μια, ένα αυτό παράδειγμα αυτό που κάνετε με τρόπο ηγετικό εξ ονόματος των πολιτών της Ευρώπης. Να πάμε στον επόμενο μιλητή τώρα και είδα στην Πρίστινα αυτό το έργο τέχνης που εγκαταστήσατε πριν τρία χρόνια Το είχα διαβάσει και το ξανακοίταξα τώρα, αλλά θα μας το εξηγήσετε φαντάζομαι. Η Αλκέτα τι έκανε. Έκανε μια έκθεση με 5.000 γυναικεία φορέματα. Θα μας εξηγήσει η Αλκέτα. Στην Πρίστινα. Για να υπενθυμίσει όλους τι συνέβη Στι γυναίκε και στα κορίτσια που ήταν θύματα σεξουαλική βία στο πόλεμο του κοσμοπεδίου. Τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για αυτά τα θέματα διεθνώ, είναι καταλληλότερη στιγμή να μιλήσει. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Οι ομιλίε δεν είναι το ένα σημείο, γιατί η τέχνη είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζομαι και ευχαρίστω να μοιραστώ μαζί σας την καλλιτεχνική μου προσέγγιση και να μιλήσω για αυτή την προσπάθεια που ονομάζεται «Σας σκεφτόμουν» και μας υπενθυμίζει τα θύματα σεξουαλικής βίας παγκοσμίω. Ξεκίνησα από το Κοσφοπέδιο, επειδή με ενέπνευσε ακριβώ, η, αυτά τα φαινόμενα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κοσφοπέδιο. Γενικά, η τέχνη μου επικεντρώνεται στην ταυτότητα, στη μνήμη και στην αλήθεια και ιδιαίτερα επικεντρώνεται στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σεξουαλική βία, κρίση προσφύγων, ισότητα φύλων και ελευθερία έκφρασης. Το πάθος μου έγκυται στην δέσμευσή μου για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δημιουργώντα λοιπόν τέχνη που ενθαρρύνει τον κόσμο να τα σκεφτεί αυτά τα θέματα, τα ενστερνίζεται και κάνει τη διαφορά. Οπτικοποιούμε αυτά που δεν μπορεί να εκφράσει κανείς. Αυτό με καθοδηγεί. Και μου δίνει μια αποστολή για την αλήθεια, για τη λύθη, για αυτό που δεν μπορεί να υποθεί, το ανίποτο και να εκφραστεί. Το 2013 ήταν μια συνέντευξη στην τηλεόραση με θύματα σεξουαλικής βίας στο Κωσυφοπαίδιο. Είδα ως γυναίκα αυτά τα άτομα αποκρίστηκαν πίσω από μια κουρτίνα ώστε να μείνουν ανώνυμα. Είπαν τι ιστορίε τους, τι προσωπικές σεξουαλικής βίας. Άκουσα να μιλάνε για το πώ το τραύμα δεν τέλειωσε αυτή την αποτρόπια πράξη, επειδή δεν είχε μόνο βιαστεί σεξουαλικά, αλλά είχε στιγματιστεί από την ίδια την κοινωνία στην οποία μεγάλωσε. Έπρεπε να ζήσει με τον φόβο της ντροπή για την οικογένειά της. τη θεωρούσαν μιας, ως μια γυναίκα χωρίς τιμή και αναγκάστηκε να μεταφέρει μαζί της ένα βαρύ αίσθημα ενοχής και τροπής χωρίς να έχει διαπράξει ποτέ κανένα έγκλημα. Ήξερα ότι δεν ήταν η μόνη. Ήξερα ότι υπήρχαν πολλές γυναίκες στο σκοτάδι, κρυμμένες που παρέμειναν σιωπηλές. Πολλές γυναίκες να από τι οικογένειε του να μην μιλήσουν για αυτή τη σεξουαλική βία στον πόλεμο, που χρησιμοποιείται ακόμα ω μέσο πολέμου και τα θύματα τη παραμένουν σιωπηλά παγκοσμίω. Μετά την συνέντευξη αυτή, κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Ήθελα οι γυναίκε αυτέ να σπάσουν τη σιωπή του, να καταπολεμήσουν το στιγματισμό και να ξέρουν ότι τη σκέφτομαι, ότι δεν είναι μόνε του. Ήξα, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα εμπλέκει όλη την κοινότητα, όχι μόνο τα θύματα. Ήθελα οι επιζήσαντες να αντιδράσουν και να δράσουν. Ήθελα να δημιουργήσω λοιπόν ένα έργο που θα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ντροπή και δεν υπάρχει στιγματισμός. Ήθελα να θέσω αυτό το ζήτημα δημοσίω σε ένα κόσμο αντρικό. Ήθελα λοιπόν να μεταφέρω αυτό το ζήτημα που δεν ήθελε κανείς να αναφέρει και να το πάω στο μεγαλύτερο γήπεδο που προσφέρουν στην Πρίστινα. Έβαλα λοιπόν αυτά τα φορέματα που κρεμάστηκαν σε, με ματαλάκια στο γήπεδο, ώστε οι φωνές αυτές να ακουστούν. Πολλές ε, γυναίκες από το Κοσμοπέδιο έδωσαν τα φορέματά τους ακριβώς για να συμμετάσχουν σε αυτή την εγκατάσταση έργου τέχνης. Συμμετέχοντας λοιπόν σε αυτή την εγκατάσταση, πηγαίνοντας στις πόλεις, συλλέγοντας τα φορέματα, μιλώντας με τα θύματα, άκουσα τις ιστορίες και ξεκίνησα ένα ταξίδι όπου οι γυναίκες μετέφεραν τις εμπειρίες τους και τις ιστορίες τους. Ήταν μια βαθιά συναισθηματικά συναισθηματική εμπειρία και επιμορφωτική για μένα και για όλους όσοι συμμετείχαν. Για πολλές από τις γυναίκες θύματα το να δώσουν τα ρούχα τους ήταν ένα είδος απε... απεμπόλησης συναισθηματικής και ενίσχυσης συναισθηματικής ταυτόχρονα. Αυτό δίνει αξία σε μεργοτέχνης. το να έχει κανείς πρόσβαση στις μάζες, να έχει ένα έργο προσβάσιμο σε όλους και όχι στους λίγους. Αυτή είναι η δύναμη της τέχνης και το τι μπορεί να πετύχει η τέχνη όταν υπάρχει μια οπτική εκπροσώπηση ανεξάρτητα γλώσσας, εθνικότητας κλπ. Αυτή η κατάσταση λοιπόν, σε σκέφτομαι, δεν αφορά μόνο το κοσμοπέδιο, αλλά τα θύματα σχολική βίας σε όλο τον κόσμο. Μιλάει μια παγκόσμια γλώσσα που μπορεί να είναι κατανοητή από όλους. Το «Σε σκέφτομαι» μας υπενθυμίζει τον πόνο και από τη φοροτιμή στις χιλιάδες θύματα που τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν έκαναν τίποτα κακό και ότι σας σκεφτόμαστε όλοι και θέλουμε να ξεπεράσετε αυτή τη σιωπή και τον στιγματισμό. Είναι λοιπόν ένα μέσο ανθρώπινης έκφρασης και αντίστασης. Μπορεί να επηρεάσει μάζες αυτό το αργοτέχνης. πέρα από τα σύνορα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι σημαντικό ανοίγει ένα ανοιχτό διάλογο με μια ποικιλομορφία φωνών και νοημάτων που ελπίζουμε θα οδηγήσουν σε κοινωνική αλλαγή. Στόχος μου ω καλλιτέχνη είναι το να μην είμαι politically correct, αλλά να είμαι αληθινή. Ως ανθρώπινο δεν μπορώ να ανεχθώ την αδικία. Δεν έχω την ε, δύναμη να κάνω πολιτικές και νόμους. Το μόνο που έχω είναι η τέχνη μου και αυτό τη χρησιμοποιώ για να αντιμετωπίσω τα πιο σημαντικά ζητήματα. Εμείς οι κοινωνικά στρατευμένοι καλλιτέχνε, αναλαμβάνουμε ρίσκα. Δεν έχουμε πόρους, πρέπει να είμαστε ερευνητές, αξιολογητές. Για να φτιάξουμε το αργοτέχνης μας πρέπει να έχουμε στήριξη πρακτική, οικονομική και θα πρέπει να εργαζόμαστε Υπό τον όρο θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, περιληπτικοί και πάντοτε ακούγοντας αυτά που έχει να μας πει ο κόσμος. Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι να παίξουμε το ρόλο που μας αντιστοιχεί, ώστε να κάνουμε διαφορά και να δημιουργήσουμε μια θετική διαφορά, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά ζητήματα όπως σεξουαλική βία. Όπως είπα πριν, χάρηκα πολύ που άκουσα φέτος ότι τον Νόμπελ Ειρήνης πήγε σε αυτά τα δύο άτομα που έκανα μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας. Και στα Δυτικά Βαλκάνια κάναμε αρκετά για να διώξουμε τους θύτες και να δικαιώσουμε τα θύματα. Δεν ξέρω. Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη, αυτό είναι κατά των ανθρωπίνων αξιών των αξιών της Ένωσης. Και ελπίζω σήμερα να έχουμε ένα κόδωνα κινδύνου για την δικαιοσύνη που χρειάζεται να ισχύσει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι δεν έχετε δύναμη, αλλά εγώ πιστεύω ότι δώσατε ένα δυνατό μήνυμα. Είναι μια απλή ιδέα στη σύλληψή της γιατί οι γυναίκε συχνά τις συνδέουμε στο μυαλό μας με απλωμένα ρούχα. Είναι ένα εξαιρετικό κόνσεπτ το κόνσεπτ που χρησιμοποίησατε. Φρικτά εγκλήματα και εύχομαι ότι οι γυναίκες αυτές ε, βρήκαν μια στιγμή ησυχία. Η σεξουαλική βία δεν είναι κάτι που, που συμβαίνει σε μέρη μακρινά, απόμακρα από τη δική μας πραγματικότητα. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στο κοσυφοπέδιο ε, άτομα που είχαν τέτοιου τύπου εμπειρίες ποτέ δεν φανταζόντουσαν ότι θα ζήσουν κάτι τέτοιο στη ζωή τους. Είναι, είναι σημάδι ότι μπορεί να συμβεί παντού και οπουδήποτε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μιλήσουν. Η Τζούλη που είναι θα θέλει να πάρει το λόγο. Είμαι πολύ συναισθηματική αυτή τη στιγμή για μια σειρά από λόγους. σπούδασα κι εγώ τέχνε πριν ε, ασχοληθώ με την πολιτική και θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η τέχνη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν ε, εξελέγην ήθελα να φέρω μία σειρά από μαρτυρίες γυναικών που είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας στη χώρα μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το, αυτή εδώ, αυτό εδώ το κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ένας χώρος που συζητάμε πολιτικές, είναι χώρος και για κουλτούρα και για τέχνη. Έχω και εγώ λοιπόν η πρώτη ε, επιτροπή στην οποία συμμετέχω είναι η Επιτροπή για τον Πολιτισμό και η Επιτροπή για τα γυναικεία δικαιώματα. Έχω εδώ φίλους μου από το Κόσοβο και πρόσφατα επισκέφτηκα τη χώρα ξανά. Πηγαίνω πολύ συχνά. Δεν πηγαίνω απλά και μόνο γιατί ε, είναι μέρος των ευθυνών μου, αλλά γιατί προσωπικά έχω δεσμευτεί απέναντι στους νέους ανθρώπους, στην κοινωνία των πολιτών, στις γυναίκες εκεί. Πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παραμένοντας δεσμευμένοι σε προσωπικό επίπεδο, όχι μόνο ως πολιτικός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να εμπλεκόμαστε σε ανθρώπινο επίπεδο, που είναι αυτό ακριβώς που έκανε το project σας. Έδωσε μια ανθρώπινη διάσταση. Γιατί πιστεύω δεν μπορούμε διαφορετικά να κάνουμε τη δουλειά μας ως νομοθέτες και πολιτικοί. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα δύο αυτά, τις δύο αυτές ταυτότητες. Πρέπει να μπορέσουμε να τις ε, χρησιμοποιήσουμε μαζί. Μπορέσαμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το κοινοβουλευτικό φόρουμ ούτω ώστε να ζητήσουμε το Κόσοβο να αποζημιώσει οικονομικά τα θύματα σεξουαλικής βίας. Και φέτος είδαμε ότι αυτό θα συμβεί. Τα άτομα λοιπόν αυτά που περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια και ξέρω ότι είναι μια διαδικασία που τραβάει σε μάκρος, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν ε, αισθάνονται άνετα όλες οι γυναίκες να κάνουν το βήμα και να μαρτυρήσουν αυτό που του συνέβη. Πιστεύω ότι τουλάχιστον βρισκόμαστε ε, στην αυγή μιας κάποιας δικαιοσύνης. Να υπάρξει δηλαδή μια νομική διαδικασία. Ήθελα απλώς δράτωμα και τις αρχές δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Με συγχωρείτε, θέλω απλά να πω ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν οι γυναίκες σε μία χώρα έχουν κάποιες εμπειρίες και κάνουν μια δημόσια δήλωση για αυτή τους την εμπειρία, ίσω μέσα από ένα έργο τέχνης ή από οτιδήποτε άλλο, παράλληλα δίνουν δύναμη και σε γυναίκες σε άλλα μέρη του κόσμου να κάνουν το, το ίδιο. Είδαμε, το είδαμε αυτό να συμβαίνει με το κίνημα Too. Οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο μίλησαν για το ίδιο θέμα. Η πορεία μου στην πολιτική έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι στην πολιτική για δικές μου προσωπικές εμπειρίες για κάτι που έζησα στην Ινδία και μου έδωσε μένα το κίνητρο να ασχοληθώ με την πολιτική. Γιατί το έκανα αυτό. Γιατί οι γυναίκες στη δική μου την κοινότητα και στο βορρά της Αγγλίας μίλησαν για κάτι που συνέβη σε μια γυναίκα σε ένα λεωφορείο στην Ινδία. Είναι πολύ δυνατές οι σχέσεις αυτές μεταξύ των γυναικών, κάτι που ε, παραδέχεται μια γυναίκα σε μια πλευρά του κόσμου, επηρεάζει γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις 17 Νοεμβρίου λοιπόν έχω ένα συνέδριο εδώ στο Κοινοβούλιο για χείρες από ολόκληρο τον κόσμο και έχω καλέσει και γυναίκες από το Κόσοβο που θα μιλήσουν και θα ανταλλάξουν τις δικές τους εμπειρίες με γυναίκες χείρες από άλλα μέρη του κόσμου που έχουν, ε, έχουν ε, πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Υπάρχει σεξουαλική βία σε πάρα πολλά μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, καλό και εσάς με χαρά, επίτροπε, αν έχετε τη δυνατότητα εκείνη την ημέρα να, να έρθετε, πείτε το σε όλους. Ελάτε να ακούσετε τις μαρτυρίες των γυναικών αυτών. Είναι θύματα σεξουαλικής βίας, έχουν χάσει τόσα πολλά πράγματα και βρίσκονται πραγματικά βρίσκονται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο και είναι ανάγκη να δείξουμε την αλληλεγγύη τους. Φέρνοντας γυναίκες λοιπόν από το Κόσοβο μπορούν να μοιραστούν τις ε, ιστορίες αυτές ε, φρικτής βίας και πιστεύω αυτό θα μας κάνει όλους μας δυνατότερους. Ευχαριστούμε την Τζούλη και για τη δική σας εμπειρία. Η Τερέσα Χιμένεθ παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα ισπανικά. Είναι το κανάλι 8, λέει η βουλευτής. Εσείς παραμείνετε στο κανάλι της γλώσσας που θέλετε να ακούσετε, γιατί αν πάτε στο κανάλι 8 θα ακούσετε ισπανικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και την, ε, το Προεδρείο γενικότερο γιατί πραγματικά βλέπω ότι όλοι κάνουν το παν για να καταπολεμήσουν τη, να καταπολεμήσουν τη βία εναντίον των γυναικών. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά και της Επιτροπής των Γυναικών, της Επιτροπής ΦΑΜ και υπάρχουν και ειδικέ ε, επιτροπές και διάφορες ε, ε, ομάδες διακοινοβουλευτικές που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω λοιπόν να απευθύνω κι εγώ έκκληση για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα εργαλείο αυτό νομικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και οδήγησε ε, στο να γίνουν πολύ πιο ορατά τα θέματα αυτά στην κοινή γνώμη. Από το δικό μας μετερίζει έχουμε κάνει πάρα πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία και για αυτή την νομοθεσία ήμουν μάλιστα προσωπικά εισηγήτρια κάτι το οποίο έχει ευνοήσει αυτόν τον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Πολλής λόγος γίνεται για την Ευρώπη. Όμως και στην Επιτροπή ΔΕΒΕ έχουμε θετήσει ψηφίσματα για να ε, καταπολεμήσουμε το βιασμό ως όπλο πολέμου. Ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα που μπορεί κανείς να διαπράξει είναι αυτό ακριβώς και γι' αυτό Χαίρομαι και αγαλιάζω όταν μαθαίνω ότι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη σε αυτούς τους δύο τόσο σημαντικούς ανθρώπους που είχαμε ε, την τύχη να γνωρίσουμε. Είναι πρόβλημα μνήμης αυτό το οποίο κάνουμε εδώ εμείς, αυτό που κάνετε εσείς με το έργο σας το καλλιτεχνικό, αυτό το οποίο γίνεται καθημερινά σε αυτό αποσκοπεί, να μην χαθεί η μνήμη, να δοθεί αυτός ο αγώνας και να νικηθεί για την αξιοπρέπεια, για τη δικαιοσύνη και για τη μνήμη των θυμάτων. Ε, οποιοδήποτε θύμα κι αν είναι αυτό Μιλούμε για θύματα τρομοκρατίας, θύματα βίας σε βάρος των γυναικών, ο, οποιοδήποτε είδους θύματα και αν είναι, πρέπει να παλέψουμε για την αξιοπρέπεια και τη μνήμη τους. Είναι αυτή η αναζήτηση της ε, αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης, γιατί η ειρήνη στο μέλλον θα, για να υπάρξει θα είναι απότοκος μόνο της δικαιοσύνης έτσι ώστε οι θήτες να πληρώσουν για αυτό που έκανα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο στο τομέα της εκπαίδευσης για να αποφύγουμε την έμφυλη βία. Πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την οτροπία έτσι ώστε οι νέοι να μην μεγαλώνουν με αυτή την οτροπία επικυριαρχίας Ξέρετε, αυτή η νοοτροπία επικυριαρχίας ξεκινάει από τη γλώσσα και αγγίζει πάρα πολλά θέματα γιατί κάνει τη γυναίκα να απεικονίζεται ως ένα πράγμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς εξού και δεν έχει, δεν έχει καμία αξία. Και γι' αυτό θα πρέπει να μπορεί η γυναίκα να εργάζεται, γιατί όταν εργάζεται είναι πιο ασφαλής, είναι πιο οικονομικά ανεξάρτητη και δεν χρειάζεται να εξαρτάται. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε από όλες, τις, ε, όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναπτυξιακή Βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ως όποιο φόρουμ και βήμα και αν σταθούμε αυτό το λάβαρο υψώνουμε πάντοτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις και να πω ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που αναφέρεται, η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Έχω μία περίπτωση όπου δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Βασνία Κρασνίφσκι είναι μία επιζώσα από το Κοσφοπέδιο. Στα 16 χρόνια, το 99 την απήγαγαν από το χωριό της και το 2014 έμαθε ότι η Σέρβια αστυνομική, ο Σέρβος αστυνομικός που τη βίασε είχε κηρυχθεί ε, ένοχος από το δικαστήριο στη Μητρόβιτσα και του είχε απονεμηθεί η ποινή της δεκαετούς ή δωδεκαετούς κάθερξης και χάρηκε διότι θεώρησε ότι απονεμήθηκε η δικαιοσύνη και αργότερα έμαθε ότι ανατράπηκε η απόφαση αυτή με την έφεση των ε, κατηγορουμένων, οι οποίοι απευθύνθηκαν και προσέφηκαν στη συνέχεια στο ανώτατο δικαστήριο. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να βελτιωθεί το δικαστικό σύστημα. Ξέρετε, είμαι μητέρα και όλοι όλοι διδάσκουμε στα παιδιά μας το ίδιο πράγμα. Προσέχετε τι κάνετε γιατί υπάρχουν συνέπειες σε αυτά που κάνετε. Πρέπει λοιπόν να είναι υπόλογοι και να λογοδοτήσουν όλοι για όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και να μην υπάρχουν τέτοιες δικαστικές ατασταλίες. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Επίτροπο, την κυρία Μυρίπα για την παρουσία τους εδώ. Να βγάλουμε μια γρήγορη φωτογραφία μαζί, αν συμφωνείτε, εδώ, με την ε, ε, με το εικονίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημαία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακριβώς από πίσω μας. Να βγάλουμε εδώ μια ε, ε, φωτογραφία στα γρήγορα, 5 λεπτά διακοπή και συνεχίζουμε στη συνέχεια.